Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, με κάποια θλίψη πρέπει να σας πω ότι είναι η τελευταία φορά κανονικά που προεδρεύω στην Επιτροπή μας και έχουμε πολύ ιδιαίτερη μέρη στη διάταξη σήμερα την ψηφοφορία για την έκθεση. Θέλω να σας ενημερώσω για την δερμηνία. Έχουμε 18 γλώσσες. Και η παρούσα συνεδρίαση, όπως και όλες οι συνεδριάσεις που είχαμε μέχρι τώρα, μεταδίδεται στο διαδίκτυο και δεν έχει έγγραφα καθόλου. Στις 2 Μαρτίου λίγη προθεσμία ε, ε, για την ε, online δημόσια πρόσκληση για στοιχεία και την υποβολή τους. Σήμερα θα ψηφίσουμε τις ε, συστάσεις και την έκθεση. Ολοκληρώνεται ένα έτος πολύ εντατικής ε, δουλειάς που ε, ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου 2016 με την συγκρότησή μας σε σώμα. Συνεδριάσαμε 27 φορές και είχαμε 47 ακροάσεις. Ακούσαμε πολλούς μάρτυρες, είχαμε και γραπτά, στοιχεία γραπτές καταθέσεις, οργανώσαμε δύο διερευνητικές αποστολές και κάναμε διάφορες μελέτες και ε, ενημερώσεις. Είναι η πρώτη ερευνητική επιτροπή, η πρώτη εξεταστική επιτροπή που ολοκληρώνει τη δουλειά της μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά γι' αυτό, αλλά τα καταφέραμε. Και σήμερα μπορούμε να ψηφίσουμε μια έκθεση πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ σαφή που πραγματικά θα κάνει τη διαφορά όχι μόνο εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά κυρίως ε, στον έξω κόσμο, τον πραγματικό κόσμο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ε, εισηγητές που έκαναν καταπληκτική δουλειά τους και τους εισηγητές και τους συντονιστές. Πρέπει να πω ότι ήταν πολύ γερή ομάδα των συντονιστών και τελικά καταφέραμε να συνεννοηθούμε και να έρθουμε σε μια κοινή γραμμή και αυτό ε, κατέστη δυνατόν μόνο με την υποστήριξη των εισηγητών, των σχεδόν εισηγητών και των συντονιστών. Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες, τους μάρτυρες που ήρθαν εδώ οι περισσότεροι και με ειλικρίνεια και με σαφήνεια κατέθεσαν βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ε, υπαλλήλους που πάντα είναι πρόθυμοι να έρχονται και να ξανάρχονται. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και το προσωπικό, διάφορε υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μα βοήθησαν, ιδιαίτερα του διερμηνεί που τι περισσότερε φορέ έμεναν και παραπάνω, 15 λεπτά μέχρι και μισή ώρα, τι υπηρεσίε ε, τη Ολομέλεια που μα έδιναν τα πρακτικά, ε, του μεταφραστέ, τη νομική υπηρεσία. Η Επιτροπή μας δεν θα μπορούσε να έχει κάνει τη δουλειά της χωρίς την νομική υπηρεσία επίσης τις ερευνητικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και ε, τελευταία, χωρίς να είναι λιγότερη σημαντική, εδώ τη γραμματεία μας και μου λένε ότι η ζωή τους θα ξαναρχίσει μόλις λήξει τις εργασίες της Επιτροπής μας. Αυτά. Έχουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης 24 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου. Ε, έχετε στα ηλεκτρονικά ντοσιέ σα. Ε, αν δεν έχετε σχόλια θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Τα σημερινά πρακτικά δεν μπορούμε πια να τα εγκρίνουμε γιατί δεν υπάρχει επόμενη συνεδρίαση. Θα διεκπεριωθεί με τη γραπτή διαδικασία αυτή η υπόθεση. Αν συμφωνείτε μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίε ευθύ αμέσω. Πρώτα το σχέδιο έκθεση. Έχω να κάνω μερικές ε, ανακοινώσεις και πάλι υπάρχει ένας ειδικό κανόνας για τις εξεταστικές επιτροπές μπορούν να ψηφίσουν μόνο τα τακτικά μέλη και οι μόνιμοι αναπληρωτές. Όσοι θέλετε να ψηφίσετε και δεν είστε τακτικά μέλη, μόνιμοι αναπληρωτέ, να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να ψηφίσετε. Ελπίζω να έχετε όλοι τι κάρτε σα, γιατί ορισμένε ψηφοφορίε ε, θα χρειαστούν έλεγχο και επαλήθευση και η τελική ψηφοφορία θα γίνει με την κάρτα. Έχουμε την απαρτία των 12 μελών που απαιτείται. Να κάνουμε μια δοκιμή για να δούμε αν λειτουργούν όλα τα μηχανήματα σωστά. Θέλετε να ξανασυμμετάσχετε στο μέλλον σε επόμενη εξεταστική επιτροπή. Αυτή είναι η ερώτηση για να ψηφίσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Η δοκιμαστική. Αρχίζει η ψηφοφορία.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 Αν έχετε προτάσεις για θέματα, ποια να είναι η επόμενη εξεταστική επιτροπή, παρακαλώ να μου τα πείτε. Λοιπόν, προχωρούμε. Ψηφίζουμε. Στην τελική έκθεση για τις μετρήσεις εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στην πρώτη παράγραφο έχουμε την τροπολογία παριθμών 8. Ψηφί πέρα παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο μάλιστα. Παρακαλώ. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 10 ψήφι πέρα Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαληθεύουμε την τροπολογία παρθμών 10 ηλεκτρονικά. Αρχίζει ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροπολογία από αριθμόν 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 15. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία Υπάρχουν 12 ψηφί υπέρ κατά. 15 is... Ε, δεν καταπίπτει, 15 απερίφθη. 12 λοιπόν υπέρ. Λέει καταπίπτει σε περίπτωση που θα εγκριθεί 15. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 13. Ψηφί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τοπολογία 14 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 16 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ, μάλιστα. Να την επαληθεύσουμε τη 17, αρχίζει η ψηφοφορία. So, closed. Απεριφθεί. Amendment 18. Who's in... Τροπολογία 18 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 22 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές Έλα. The vote is open. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας. Προχωρούμε συμβαστική 2. Ψηφί πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να την ελέγξουμε. Θέλετε τη συμβαστική 2, ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα. The vote is closed. That is accepted. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 ως προσθήκη θα τη ψηφίσουμε. Ψήφι Κατά. Αποχές. Rejected. Απορρίπτεται. Πάμε στην 33. Ψήφι Κατά. Έλεγχος. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Ψήφι Κατά. Δεν είναι σαφές. Έλεγχος. Μέσα στην τροπολογία 36. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία αριθμό, 31. Ψηφί Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Αρχίζει τώρα. Για την τροπολογία 35. Πέρασμα. Απορρίπτεται. Η 32 ψήφι Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 ειπε Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 7, 40, έχουμε προφορική τροπολογία. Τη γνωρίζετε όλοι. Ωραία, ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά στο τσακάρουμε αρχίζει η ψηφοφορία. Και τελειώνει. Εγκρίνεται σαφέστατα. Λοιπόν, συμβαστική 14. Ψήφι Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Ψήφι Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κάτι λάθος θα έκανα, αλλά στο ελέγξουμε για να το λέτε. Αρχίζει ψηφοφορία. Closed. <laughs> Okay. That is Ναι. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τσεκ για τη 49. Πάμε. Αρχίζει και τελειώνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 50. Who's in favor? 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 και 53 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. We move to 59 parts. 59. Στο δεύτερο τμήμα όμως. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. έχουμε λοιπόν 59 τμήμα δεύτερο. Αρχίζει ψηφοφορία. Vote is closed. That is accepted. Πέρας εγκρίνεται. 62. Who's in favor? 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Against. Κατά. Έλεγχος. Αρχίζει τώρα. Στην τροπολογία 64. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Για 77 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Στην 80. Αρχής. The vote is closed. That is rejected. Πέρας απορρίφτεται. We move to compromise 4. Ε, συμβαστική 4. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ 88 είμαστε υπέρ κατά απορρίπτεται. Α, αποχές ξέχασα. Απορρίπτεται. Έλεγχο θέλετε για την 88. 88. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. is... Πέρας. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. against? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά απόχες νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά αφού είναι συμβιβαστική καλύτερα να την ελέγξουμε πάμε αρχίζει λοιπόν η επαλήθευση στην 13 Περισσεύει ένας φιλελεύθερος, λυπάμαι πάρα πολύ. Απορρίπτεται. 93 είπε. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 94 είπε. Κατά. Αποχές. Δεν ήταν πάρα πολύ σαφές. για το ελέγξουμε. Ψηφίσουμε λοιπόν την 94. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα, στην 95 έχουμε τμήματα. Ε, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. Πέρα, ε, ε, ε ένταξη της Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. 95 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 97. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Την 97. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Διαθετείτε. 105. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Την 105 με ψηφοφορία. ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην 106 και 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 111. Υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Κατά. εποχές Υιοθετείται. 116. Υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 121 υπέρ.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 Ελέγχουμε την 130 ηλεκτρονικά. Πέρας προφορίες. Υιοθετείτε. Εκατόν τριάντα δύο υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά απο... αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά Εποχές. απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Εποχές. απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε τώρα. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 144 και 145 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Εποχέ Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Εποχές Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Εποχές Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Εποχές Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε την 158. Ψηφίσετε. Πέρες ψηφοφορίας. Προφανώς απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. Συμβασμός 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. Συμβασμός 8 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 171 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 175 υπέρ, όχι, διορθώνει 174, διορθώνει πρόεδρος, 174 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 175 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται, 178 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τσεκ. Ελέγχουμε την 178 ηλεκτρονικά. Αν μπορείτε να ρωτήσω κάτι. Να ψηφίσουμε την τροπολογία 174. Γιατί δεν θυμάμαι τώρα αν εγκρίθηκε. Θέλετε να ελέγξουμε την 174, έτσι. Λοιπόν, ελέγχουμε την 174 με ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία της 178. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 178 τώρα. Πέρσι Υιοθετείτε. Τώρα πάμε στην 180. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 185 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι υιοθετείται, αλλά στο ελέγξουμε. Σφίσουμε τώρα. Πέρες φοφορίας. Υιοθετείται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 187 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 191 τώρα. ψηφοφορίας απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 194 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 194. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας οφορία. Κατόν 195 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές Ελάτε, πάλι τα ίδια. Ηλεκτρονικό έλεγχο. Οι μισοί δεν ψηφίζουν καν. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα την 198 ηλεκτρονικά. Θα το ξανακάνουμε. Ξαναψηφίζουμε την 198.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 Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 3. Υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, πρέπει να το ελέγξουμε. Ψηφίσετε τώρα. Την 6. Πέρες ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Ούτως ώστε να δουν οι πολιτικές ομάδες τι αποτελέσματα είχαμε. Συνάδελφοι, είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Δεν αφορά μόνο το σύνολο, αλλά και τα, ε, Και τα πραγματικά περιστατικά. Μια νέα ψήφος και για τα δύο δηλαδή. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. And the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. συγχαρητήρια στους εισηγητές, να τους ενημερώσω μόνο ότι δεν ψήφισα, γιατί έχω πλήρη εκπροσώπηση από την ομάδα μου. Αλλά είναι ότι θα ψήφιζα υπέρ. Λοιπόν, προχωράμε στη δεύτερη έκθεση του σχεδίου συστάσεων εν συνεχεία της έρευνα σχετικά με τι μετρήσει των εκπομπών στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανία. Ξεκινάμε με τη συμβαστική 1 υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείτε. Οι 11 και οι 12 είναι ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, 10 και 11, συγγνώμη, είναι ταυτόσιμες, απορρίπτεται, οι 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στη 12, άρχεται η ψηφορία. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά να ελέγξουμε συμβαστική 11. Συγγνώμη. The vote is closed. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται συμβαστική ενέα. Θέλετε να αλλάξουμε την 21, λοιπόν, ψηφίζουμε. And the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίζει την 29 και απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική ενέα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 35, 36, συγγνώμη, υπέρ, κατά και εγκρίνεται. Περνάμε στην 37, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία 39, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται Σαράντα. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για 39. Πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Um, Σαράντα. Υπέρ. δεν ψηφίζουμε γιατί έχουμε πλήρη εκπροσώπηση από την ομάδα. Στις 40 λοιπόν, υπέρ κατά. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε τη 40. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά. αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα την ελέγξουμε και αυτήν την 52 ανοίγει η ψηφοφορία The vote Πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά. Θα ψηφίσουμε στην συμβαστική 10. Ανοίγει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Περνάμε στην 58. Υπέρ. Κατά αποχές και απορρίπτεται 61 υπέρ κατά δεν είναι σαφές θα αλλάξουμε πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται πάμε στην 62 τμήμα 1 υπέρ κατά ελέγχουμε την 62 ε, τμήμα 1 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Περνάμε στην 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά ελέγχουμε. Ανοίγει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και ξεκάθαρα απορρίπτεται η 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 27 86 συγγνώμη και 87 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 και 90 και 91 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά θα ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ 96 94 είμαστε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές και απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε την 96, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 ψηφορεί σε τμήματα, τμήμα 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα 2, υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε το τμήμα 2 της 99. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 100, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 101 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε την 104, λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 109 και 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 και 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ήταν τόσο σαφές, γιατί ψήφισαν διαφορετικά οι ομάδες, σας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 115 και 116 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Ανοίγει η ψηφορία. Πέρας. Όχι ακόμα. Τώρα. Και απορρίπτεται. Περνάμε στην 120 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 122. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πολλοί όμως δεν σηκώνουν το χέρι και γι' αυτό είναι δύσκολο να δω. Λίγες σελίδες μας μείνανε και τελειώνουμε. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 126-127 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Και με αποχές, εντάξει. Αποχές. Α, τώρα θέλει έλεγχο όμως. 128 Εγκρίθηκε. 130 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 131. Όχι, 129 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Στην 132. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Δεν είναι πολύ σαφή τα πράγματα, ας τα ελέγξουμε. 137 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Δεν κρίνεται. 138 Πε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 139 και 140 ψήφι πε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 147 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έχουμε μια προφορική τροπολογία εδώ της κυρίας Βονταλόν Μπονφουά. Συμφωνείτε όλοι να ψηφίσουμε την προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 σε δύο τμήματα τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές ε, αυτό θέλει έλεγχο αρχίζει η ψηφοφορία πέρας Απερίφθη. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 175 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται εγκρίνεται διορθώνει η πρόεδρος 176 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 177 υπέρ κατά, αποχές απορρίψεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές απορρίψεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε λοιπόν την 178, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Τώρα απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία είναι 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Οι δύο, σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. κατά, αποχές. Adopted. Okay. No, let's not go wrong here. Εγκρίνεται. Κάτσε μην κάνω κανένα λάθος. Βήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. έλεγχο, γιατί δεν είναι σαφέ. Παλτεύουμε την 4 αρχή τώρα ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Τροπολογία παρθμών 3 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 υπέρ. Κατά χέρι εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στη τελική ψηφοφορία. Ζητάει κανείς διάλειμμα? Όχι. Ωραία, ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας κρίνεται, θαυμάσιο το αποτέλεσμα, πολύ μεγάλη πλειοψηφία και πάρα πολλά συγχαρητήρια επίσης στους εισηγητές μας, στους σκιώδεις, σε όλους εσάς. Αν δεν έχουμε τίποτα άλλο, θα τα ξαναπούμε στην Ολομέλεια. Και σας υπόσχομαι ε, ότι θα το γιορτάσουμε κιόλα, κάτι θα πιούμε. Ήταν πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα στην Εξεταστική μας Επιτροπή και καλή τύχη για την Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ.